Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρακαλώ, καθίστε. Κυρίσω την έναρξη της περίοδου Συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και διακοπής της 24 Μαΐου του 2012. Τα πρακτικά